Ε, Παρακαλώ, καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μία συνεδρίαση αρκετά μακροσκελή με πολλές τοποθετήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να μην περιμένουμε πολύ για να αρχίσει η συνεδρίαση. Καλωσορίζω όλους σας αυτήν την ε, κοινή συνεδρίαση. Θα βλέπετε στο Προεδρείο, είναι η συνάδελφος Ζολή, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, η συνάδελφος Χάουταλα, η οποία είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε ως προσκεκλημένους εδώ και τα μέλη των αντιστοίχων επιτροπών. Όπως γνωρίζετε με την τωρινή συζήτηση ξεκινάει η διαδικασία για την ε, απονομή του βραβείου Ζαχάροφ για το 2010. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ε, διαδικασία που ξεκίνησε το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βραβείο αυτό αναγνωρίζει το έργο ανθρώπων, ε, μεμονωμένων ανθρώπων ή οργανώσεων οι οποίοι με κίνδυνο της ζωή τους πολλές φορές ε, στρατεύονται για να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ανοχή, την ελευθερία. και αντιστέκονται στην ε, κατά πίεση και την ε, παραβίαση όλων αυτών των δικαιωμάτων. Στο βραβείο δόθηκε το όνομα της μεγάλης προσωπικότητας, του μεγάλου φυσικού που συνεπεί σε αυτές τις αρχές πάλεψε όλη τη ζωή. Η τελική απόφαση είναι μια απόφαση της διάσκεψης ε, των προέδρων των ομάδων, αλλά εμείς σήμερα με τη συζήτηση που θα γίνει και με την ψηφοφορία στις 18 του μηνός στο Στρασβούργο συμμετέχουμε ένεργα στην ε, διαδικασία επιλογής όπως επίσης με τη δημοκρατική συζήτηση που γίνεται προσδίδουμε νομιμότητα και δημοκρατικότητα σε αυτή την απόφαση. Συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να παραμείνω κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας εύχομαι καλή δουλειά και είμαι ιδιαίτερα αλληλέγγυος μαζί σας. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο Χάουταλα η οποία θα προεδρεύσει των εργασιών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη. Εγώ θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το πέρας της προθεσμίας, το πέρας της προθεσμίας 22 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, διορία δηλαδή για την υποβολή υποψηφιότητων, η γραμματεία είχε λάβει 9 υποψηφιότητες και η γραμματεία εξετάζει, ε, μάλλον θεωρεί ότι είναι όλες αποδεκτές όσον αφορά το καθεστώς που διέπει την απονομή του βραβείου. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να βρείτε περιγραφές όλων των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένου ενός σύντομου βιογραφικού στους φακέλους σας. Οπότε ρίξτε μια μάτια, παρακαλώ. Και επίσης ε, σύντομα να παραθμίσω τους εννέα υποψηφίους και έπειτα να δώσω το λόγο ένα προς ένα σε ένα μέλος που θα παρουσιάσει το συγκεκριμένο κάθε φορά υποψήφιο καθένα θα έχει έξι λεπτά στη θέση του. Μπορώ να δείξω κάποια ευελιξία για σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν πάνω από ένα που θέλουν να παρουσιάσουν τον υποψήφιο του. Ελπίζω πως, ωστόσο πω κανένα δεν θα υπερβεί το όριο των 6 λεπτών ανά υποψήφιο. Διότι πρέπει να επικρατήσει ισότητα για του υποψήφιου, να έχουν δηλαδή ίσε ευκαιρίε για να παρουσιαστούν σε αυτή τη συνεδρίαση. Καταρχήν, λοιπόν, με αλφαβητική σειρά έχουμε το ε, κίνημα πολιτών Access Έχουμε τον κύριο Χάιταμ Αλμαλέ, Breaking the Silence, Γιγέρμο Φαρίνιας, εξ ονόματος όλων όσων αγωνίζονται για την ελευθερία και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, Αμινέτου Χαϊντάρ, Ντάβιτ Ισακ, η κυρία Μπερτουκάν Μιτέξα, Πατήρ Γκουγέν Φανλή, και έχουμε και την αποστολή Open Doors. Θα σας ε, τους παρουσιάσουν οι υποστηρικτές τους που θα περιγράψουν τους διάφορες δραστηριότητε τους και η παρουσίαση γίνεται και πάλι με αλφαβητική σειρά. Παρακαλώ να μην υπερβείτε λοιπόν το όριο των 6 λεπτών, ακόμα και αν είστε πολλοί που θα παρουσιάσετε τον κάθε υποψήφιο. Καταρχήν λοιπόν να καλέσω και κυρία Σάκη να παρουσιάσει την οργάνωση Access. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κίνημα πολιτών ε, Access είναι ένα κίνημα το οποίο ε, υποστηρίζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι ένα κίνημα το οποίο βοηθά στην ε, κρίσιμη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κίνηση προς την ε, ελευθερία και όχι στη λογοκρισία, ή σε δικαιώματα στο ψηφιακό μέλλον. Η άξες δημιουργεί ένα δρόμο όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν στο ανοιχτό ίντερνετ παρά την ε, εποπτεία ή καταπιστικά καθεστώτα κατά πολιτών που εμποδίζουν εκατομμύρια ανθρώπων να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ σήμερα. Στόχος είναι δηλαδή να υπάρχει αυξημένη ασφάλεια και ποιότητα χωρίς ε, όμως φόβο ή έλλειψη. Θέλει να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών και τις ε, μειονότητες να μπορέσουν να συμμετέχουν δίνοντας ε, πολιτικές συμβολές σε αυτή τη νέα, τη νέα μορφή υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων online. Ε, δημιουργούν ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτών που υποστηρίζει αυτούς τους στόχους. Η Access δημιουργήθηκε μετά από το κίνημα μετά, που δημιουργήθηκε μετά από την καταστολή στο Ιράν των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ η Άξες έδωσε κρίσιμη τεχνική υποστήριξη που βοήθησε να μείνει ανοιχτό το ίντερνετ για το δημοκρατικό κίνημα του Ιράν. Και καθώς εκατομμύρια αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα των εκλογών, οι ακτιβιστές μπόρεσαν online ε, να διατηρήσουν διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το, αλλά και διάφορα blog και διάφοροι ιστότοποι ανοιχτοί. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές χώρες όπου ο κόσμος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα έχουν βοηθήσει να απελευθερωθούν χιλιάδες βίντεο διαμαρτυρίες αλλά και ε, κατάχρηση ανθρωπίνων και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα είδαν εκατομμύρια άνθρωποι online. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες με βίντεο σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ξεπεράσουν ε, το, τους φραγμούς, να φτάσουν σε συγκεκριμένες ιστότοπους αλλά και να ειδοποιήσουν τις ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τις απαγορεύσεις και τους φραγμούς των ε, πολιταρχικών καθεστώτων. Ε, η Άξης βοήθησε και ε, στη, στο Ιράν. Ε, ε, ε, λειτουργεί λοιπόν για την προστασία και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια ομάδα ψηφιακής βοήθειας που μπορεί να αναπτύξει τεχνολογίες κατά της εποπτείας, κατά των φραγμών και κατά της λογοκρισίας. Επίσης δημιουργούν ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτών όπου μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί να βοηθήσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και να προωθήσει την ψηφιακή ελευθερία. Αλλά επίσης έχουν δημιουργήσει ένα κέντρο μέσων μαζικής ενημέρωσης για να ενημερώσουν τον κόσμο όπως ε, και εμάς ε, για το τι διακυβεύεται ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω του ίντερνετ. Σχεδόν 4 στους 5 ανθρώπους ολόκληρο τον κόσμο και φτάνει να θυμηθεί κανείς πόσος κόσμος ε, είναι νεότερος κάτω των 30 ετών και για αυτούς η πρόσβαση στο ίντερνετ έχει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Τέσσερι στου πέντε λοιπόν πιστεύουν πω η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι ένα θεμελιώδε ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά πάνω από το 30% του κόσμου ζει σε κατάσταση λογοκρισία και απειλή όσον αφορά τη χρήση αυτή τη τεχνολογία. Η πρόσβαση στο ίντερνετ όχι μόνο είναι λοιπόν δικαίωμα, είναι και μια πύλη όσον αφορά άλλα δικαιώματα όπως η, έκφραση, η ελεύθερη έκφραση, η η μεταχείριση, η πρόσβαση στην ενημέρωση και ούτω καθεξής. Στο Ιράν επίσης δολοφονήθηκε μια νέα και πολλά υψχόμενη κοπέλα η οποία πυροβολήθηκε επειδή εκφράστηκε ελεύθερα. Αυτό το μαγνητοσκόπησε ένα κινητό τηλέφωνο και μετά διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ ε, και έτσι δημιουργήθηκε παγκόσμια κατακραυγή. Νομίζω πως ε, είναι κατανοητή η σημασία των ε, πληροφοριών της επικοινωνίας σήμερα. Μπορεί κάποιος να βασανιστεί όσον αφορά το κωδικό τους για το, το προσωπικό λογαριασμό email. Βλέπουμε να παρακολουθούνται κινητά τηλέφωνα και να φυλακίζονται και διάφοροι που λόγω και, μόνο και μόνο επειδή έχουν blog και, και εκεί μιλούν ελεύθερα και εκφράζουν την άποψή τους. Στο Ιράν έχουν φυλακιστεί άνθρωποι για αυτό το λόγο. Να σας θυμίσω διάφορες χώρες όπου οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να λογοκρίνουν τον κόσμο. Μιλήσαμε για το Ιράν, αλλά επίσης συμβαίνει στην Αίγυπτο που φυλακίζονται οι bloggers και στο Αζερβαϊτζάν και η Κίνα ασκεί ένα καταπιεστικό τέτοιο καθεστώς, η Βενεζουέλα, η Βυρμανία, η Κούβα και πολλές άλλες χώρες. Η Χίλαρη Κλίντον ε, έβγαλε ε, μια ομιλία υπογραμμίζοντας ε, το ρόλο που παίζουν οι νέες τεχνολογίες στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ελεύθερη έκφραση. Νομίζω λοιπόν πως η Access είναι μια οργάνωση εξαιρετική και πολύ καλή υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ. Σας ευχαριστώ πολύ και να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι υπάρχει ένα βίντεο που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σας δείξουμε εδώ. Δεν ξέρω ξέρω αν να κάνουμε λογοκρισία, αλλά φαντάζομαι πως όλοι θα μπορέσετε να το δείτε, να δείτε ποια είναι η ιστορία της άξης και ποια είναι η ιστορία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βοηθήθηκαν από την τεχνολογία αυτή της οργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ε, υποψήφιος είναι ο κύριος Χάιτα Μαλμαλέχα, με τα καταλφαβητική σειρά. Και επειδή εγώ είμαι η πρώτη προσυπογράφουσα για την υποψηφιότητά του, θα ζητήσω από τον κύριο Τόνσκης να παρουσιάσει την υποψηφιότητα. Είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι ευχαριστησή κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, να περιγράψω τον κύριο Σίρναλ Αλμαλέχ, Σύριο δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτάθηκε από την κυρία Χάουταλα και άλλους συναδέλφους. Ένα έτος μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος για τον Μοχάμετ Αλχασάνη, ένα Σύριο δικηγόρο ο οποίος συνελήφθη αυθαίρετα και κρατείται στην απομόνωση, το Σεπτέμβριο φέτος υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Συρία με ειδική αναφορά στην υπόθεση του Χαϊτά ενό ενός 80χρονου δικηγόρου υπηρεσίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Χαϊτά Μαλμαλέ συνελήφθη αυθαίρετα από υπαλλήλου γενική υπηρεσία Πληροφοριών στι 14 Οκτωβρίου 2009 κρατήθηκε σε απομόνωση ω την ανάκρισή του από στρατιωτικό εισαγγελέα στι 20 Οκτωβρίου του 2009 και δικάστηκε από το δεύτερο στρατοδικείο τη Δεμαρκού παρά το γεγονός ότι τα στρατοδικεία δεν μπορούν βεβαίω να δικάσουν πολίτες. Η σύλληψή του έλαβε χώρα την περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη πρότειναν να υπογραφεί συμφωνία σύνδεση με τη Συρία, στην οποία βεβαίω υπάρχει και ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 4 Ιουλίου 2010 ο Χαϊτά Μαλμαλέ καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων και υπερβολικών ειδήσεων που αποδυναμώνουν το εθνικό φρόνημα βάσει των άρθρων 285 και 286 του ποινικού κώδικα της Συρίας. Οι κατηγορίες προκύπτουν από τις συνεντεύξεις του κυρίου Αλμαλέ στα ΜΜΕ, στις οποίες επέκρινε τη συνεχιζόμενη χρήση αναγκαστικών νόμων στη Συρία και τον συνεχιζόμενο έλεγχο των αρθών της χώρας στο δικαστικό σύστημα. Ε, Αποστολέ παρακολούθηση τη δίκη που οργανώθηκαν από διεθνεί οργανώσει κοινωνία των πολιτών ανέφεραν ρητά ότι η δίκη του κυρίου Αλμαλέ δεν πληρούσε τα διεθνή πρότυπα δίκαιη δίκη. Η υγεία του κυρίου έχει επιδεινώθηκε σοβαρά το καλοκαίρι, πάσχει από αρθρίτιδα, διαβήτη και προβλήματα του θηριοειδού και δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά του. Η καταδίκη του Χαϊτάμ Αλμαλέχ, ο οποίο θεωρείται εξέχων δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδεικνύει τι συγχυνόμενες διώξει δικηγόρων και υπραστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνιστά επίση μια έντονη προειδοποίηση προς τους δικηγόρους που προάγουν το κράτος δικαίου και αμφισβητούν καθημερινά του περιορισμούς που επιβάλλει η κατάσταση εκτάκτης ανάγκη, η οποία ισχύει από το 1963. Η υπογραφή σύνδεσης Ένωσης Συρίας καθυστέρησε ύστερα από έτοιμα τη Συριακής πλευράς. Από τον Οκτώβριο του 2009 η Επιτροπή έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να βρει έναν τρόπο για την υπογραφή της συμφωνίας. Στο ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 2010 το Κοινοβούλιο υπογράμμισε την επιδείνωση κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένη συστηματική καταστολή σε βάρο δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και ζήτησε τη θέσπιση ενό σαφού μηχανισμού για την έναρξη συζητήσεων μεταξύ των Σύριων και Ευρωπαίων εταίρων σχετικά με τι συγκεκριμένε βελτιώσει των μισών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία που αναμένει η Ένωση από τι αρχέ τη Συρία η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ του 2010 στον κύριο Αλμαλέχ θα μπορούσε να εκλειφθεί ως σημαντική υποστήριξη όλων εκείνων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη Συρία και θα αποτελούσε ένα σημαντικό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να διασφαλίσει συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα τη εξωτερική δράση τη όσον αφορά το σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί προσωπικού την ευχαρίστηση να οργανώσω ένα σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τονίσουμε την κατάσταση του κυρίου Αλμαλέχ. Και συμμετείχε και ο ιός το οποίος είναι δικηγόρος. Το σεμινάριο αυτό λοιπόν με οδήγησε στο συμπέρασμα πως ο κύριος Αλμαλέχ Σύριο πατριώτη και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξίζει πραγματικά το βραβείο Ζαχάροφ 2010. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόνσκης. Δεν ανέφερα πως η Access προτείνεται από, ε, από τους φιλελεύθερους και ο κύριος ε, Αλμαλέχ από εμένα και άλλους 44 συναδέλφους. Λοιπόν, φτάνουμε στον τρίτο υποψήφιο με αλφαβητική σειρά που προτείνεται από τους πράσινους και την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και την παρουσίαση θα κάνει ο Ντανιέλ Κονμπεντίτ. Και για την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θα μιλήσει η Μαρή Κριστίν Βερζιά. Κύριε Κονμπεντίτ, έχετε τον λόγο. Merci. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω το ρήγμα στη σιωπή, το Breaking the Silence, δεν αποτελεί επιχείρημα κατά των άλλων υποψηφίων. Όλοι οι άλλοι υποψήφοι είναι υποψήφοι και υποψήφιες άξιοι για το βραβείο Ζαχάροφ. Αυτό είναι σίγουρο προτείνουμε την Breaking the Silence για έναν απλό ε, λόγο. Στην ε, περιοχή Ισραήλ-Παλαιστίνης σήμερα παίζεται το μέλλον των δύο λαών. Παίζεται ο πόλεμος και η ειρήνη. Διότι αν αυτές οι διαπραγματεύτες οι οποίες ξεκίνησαν, οι οποίες είναι τόσο επίπονες, σταματούσαν λόγω της επέκτασης της κατοχής και των επικισμών τόσο εκ μέρους του Ισραηλινού στρατού αλλά και λόγω της τάσης ορισμένων Ισραηλινών πολιτών δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η ιστορία σε εκείνη την περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεράστια ευθύνη για το τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περιοχή. Η ομάδα Breaking the Silence, η οποία αποτελείται από Ισραηλινούς στρατιώτες που έκαναν τη θητεία τους, υπηρέτησαν τη θητεία τους στα κατεχόμενα εδάφη, η πρώτη στη Χευρώνα κατά την πρώτη τυφάδα και ή άλλοι στην ε, στρατιωτική παρεπέμβαση στη Γάζα. Είναι στρατιώτες που καταμαρτυρούν για την παρανομία ορισμένων πράξεων του Ισραηλινού στρατού. Δεν αμφισβητούμε την Ισραηλινή δημοκρατία. Αλλά η ιστορία απέδειξε δημοκρατικές χώρες όταν κατέχουν άλλες χώρες εγκαταλείπουν τη δημοκρασία. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Γαλλία όταν κατήχε την Αλγερία. Η Γαλλία ήταν μια δημοκρατία αλλά ο γαλλικός στρατός στην Αλγερία ε, ε, λειτουργούσε αντιδημοκρατικά γιατί ήταν ένα στρατός κατοχής. Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατό κατοχής στην περιοχή. Μιλάμε λοιπόν για την Breaking the Silence, την, την υπερασπιζόμαστε γιατί πρόκειται για θαραλέους άντρες και γυναίκες οι οποίοι επέλεξαν την απομόνωση τελικά, διότι τους απομονώνει η Ισραηλινή κοινωνία. Δεν θέλει η Ισραηλινή κοινωνία να ακούει για την πραγματικότητα της κατοχής. Σας καλώ όλους. Πάτε να δείτε τη Χευρών. Δείτε τι είναι η Χευρών. 350 Ισραηλινοί έπικοι, συν μία γεσιβά, δηλαδή μία θρησκευτική σχολή, καταπιέζουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες Παλαιστινίους. Δηλαδή 300 Ισραηλινοί ε, και ε, ε, μεταχειρίζονται τους Παλαιστινίους με έναν φρικτό τρόπο. Και ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει αυτή την κατοχή της Χευρών. Όταν ψηφίζουμε, προτείνουμε την Breaking the Silence, ψηφίζουμε για την ειρήνη, ψηφίζουμε για την τιμή της δημοκρατίας του Ισραήλ. Όταν ψηφίζουμε την Break the Silence λέμε θέλουμε δύο κράτη, ένα Παλαιστινιακό και ένα Ισραηλινό και υπερασπιζόμαστε τους ειρηνιστές όλων των πλευρών, ειρηνιστές Παλαιστίνιους και ειρηνιστές Ισραηλινούς που αποτελούν την τιμή και την ευκαιρία της ειρήνης. Εμείς παρεμβαίνοντας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να δώσουμε μία ευκαιρία στην ειρήνη. Give peace a chance. Λοιπόν, breaking the silence. Λοιπόν, ας δώσουμε μία ευκαιρία στην ειρήνη και ας ψηφίσουμε την breaking the silence. Ας πάσουμε τη σιωπή. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο για να παρουσιάσει το δικό της υποψήφιο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Κον Μπεντίτε. Θα εξηγήσω λίγο πιο τεχνικά το τι είναι η Breaking the Silence. Είναι μια ένωση που συγκροτήθηκε το 2004 για να μπορέσει να δώσει το λόγο στους Ισραηλινούς στρατιώτες που γύριζαν στα σπίτια τους και που πραγματικά ήταν μπλοκαρισμένοι από τη σιωπή, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Αυτή η Ένωση μάζεψε μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, για επεισόδια για τα οποία ήταν μάρτυρες αυτοί οι στρατιώτες, ε, για πρακτικές που άσκησαν αυτοί οι στρατιώτες ε, κατά Παλαιστινίων πολιτών, αμάχων. Αυτή η Ένωση λοιπόν κοινοποιεί αυτή την αλήθεια στο Ισραήλ, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή την Ένωση την υποστηρίζουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση την οποία επέκρινε η Ισραηλινή κυβέρνηση θεωρώντας απαράδεκτο να χρηματοδοτούμε ενώσεις σε μια δημοκρατική χώρα και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να πάνε να δούνε τι γίνεται στις τρίτες χώρες. Αυτά μας είπε η κυβέρνηση. Αυτά τα λέει επιλέξει. Η Breaking the Silence συνέχισε τη δουλειά της. Έχουμε πολλές από τις μαρτυρίες της Breaking the Silence στην έκθεση Goldstone. Άμα δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες της Breaking the Silence, η έκθεση Goldstone δεν θα είχε αυτή τη δύναμη που έχει. Πρόκειται για μία ένωση η οποία απειλείται από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η εκστρατεία που η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει την Breaking the Silence. Όπως είπε ο πρόκειται για ένα σύμβολο για το τι συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και όπως λέμε πάντα κυρία Πρόεδρε, τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να είναι τα ίδια παντού και για όλους. Ευχαριστώ. Περνάμε στον τέταρτο υποψήφιο με αλφαβητική σειρά, τον κύριο Γκυγέρμο Φαρίνες. Εξ ονόματος ε, όλων όσων αγωνίζονται για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα. Και τον έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Χριστιανοδημοκράτες, και η Ευρωπαϊκή Συντηρητική και Μεταρρυθμιτές και ο Έντιβαρτ Κοζούσνικ και 91 άλλοι. Το πρώτο μέρος παρουσίασης θα το κάνει ο Ιγνάσιος Αλαφράνκα, ο Σάριος Βόλσκι και ο Βαρανέσσα και το δεύτερο μέρος ο κύριος Κοζούσνικ. Σας παρακαλώ να λάβετε επίσης υπόψη το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, δύσκολα μπορεί κανείς να βρει υποψήφιο που να ανταποκρίνεται απόλυτα στο προφίλ του βραβείου Ζαχάροφ όσο ο Γιγέρμο Φαρίνας. Είναι ψυχολόγος, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα τον τίμησαν με το βραβείο τους και επέλεξε την παθητική αντίσταση στην Κούβα. Στις 4 Φεβρουαρίου φέτος ξεκίνησε απεργία πείνας. Όχι υπέρ του ιδίου, αλλά για την αλληλεγγύη των 24 συντρόφων του. Και μετά από μεσολάβηση ε, της ε, Καθολικής Εκκλησίας της Κούβας αποφυλακίστηκαν οι συγκρατούμενοι του. Υποφέρει αυτός ο άνθρωπος από τις 23 απεργίες πείνας που έχει κάνει. Βέβαια η πείνα δυνάτησε το κορμί του αλλά όχι το πνεύμα του. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένας αξιοπρεπέστατος υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ κύριο Σάουρος Βόλσκι είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Φαρίνιας είναι ένας, ένας εμβληματικός αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγωνιστής χωρίς ε, τη βία και προτείνουμε να του δοθεί αυτό το βραβείο εξ ονόματος των ε, αγωνιστών της ελευθερίας της Κούβας. Είναι νομίζω αυτονόητη η υποψηφιότητά του. Ανταμείβουμε διάφορους αγωνιστές της ελευθερίας που έχουν πληρώσει διάφορα τιμήματα φυλάκισης ή θανάτου ακόμη. Εδώ όμως είναι ένας εξαιρετικό, εξ, εξαιρετικός υποψήφιος ε, με πολιτική συνείδηση. Αποφάσισε 23 φορές να κάνει απεργία πείνας, να ρισκάρει τη ζωή του για να απελευθερωθούν πολιτικοί κρατούμενοι και να αλλάξει έστω και λίγο το καθεστώς του Κάστρο. Είναι μια υποψηφιότητα που νομίζω ότι σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο πλήρει όλα τα κριτήρια που θέτουμε όταν θέλουμε να ανταμείψουμε τους ανθρώπους με το βραβείο Ζαχάροφ. Γι' αυτό και πλήρως και με όλη μας την καρδία υποστηρίζουμε αυτή την υποψηφιότητα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάιρους Βόλσκι. Τώρα ο Γιάννος Λαβαλέσα. Σας ευχαριστώ. Αυτό το βραβείο είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Ευρωκοινοβούλιο να τονίσει και να δείξει όχι μόνο τη ζωή ενός ανθρώπου αλλά και τις αλλαγές που γίνονται μέσα σε μια κατάσταση. Είναι δύσκολο ακόμα να πούμε ότι θα αλλάξει το καθεστώς στην Κούβα αλλά βλέπουμε πως το σύστημα, το κουβανικό καθεστώς αρχίζει να καταραίει και πιστεύω πως η αξία του κυρίου Φαρίνιας που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς συμβολίζει την ίδια την ιδέα του βραβείου Ζαχάροφ. Το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε δηλαδή βραβεύοντάς τον να δώσει ένα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό μήνυμα κατά της έλλειψης σεβασμού, κατά της έλλειψης ε, ελευθερίας στην Κούβα, κατά της ε, απάνθρωπης μεταχείρισης των πολιτικών κρατουμένων, αλλά και να στηρίξει τη μελλοντική ε, πολιτική σκηνή στην Κούβα. Ο κύριος Κοζούσνικ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το βραβείο Ζαχάροφ είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ίδιος ο Ζαχάροφ όταν το 1968 κατέλαβαν τη χώρα μας τα στρατεύματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο Ζαχάροφ ήταν ένας από τους λίγους που μίλησαν. Θα μπορούσε να έχει μία ίσχυη ζωή ενός σοβιετικού επιστήμονα ή τη ζωή ενός ε, αντιφρονούντα και δεν δίστασε στιγμή να διαλέξει. Πρέπει λοιπόν να τιμούμε ανθρώπους σαν τον Ζαχάροφ. Όταν ο Ορλάντα το Μάιο πέθανε σε μια κουβανική φυλακή, ένας άλλος άνθρωπος, ο Γιγέρμο Φαρίνιας, ε, τον υπερασπίστηκε και η δική του η υγεία υπέφερε από την απεργία πίνες. Δεν δίστασε όμως ούτε και αυτός ε, στιγμή να αγωνιστεί για την ελευθερία της ε, Κούβας. Η ζωή του είναι παρόμοια με την ζωή του Ζαχάροφ και βεβαίως η Κούβα ακόμα αναμένει την ελευθερία. Ο κύριος Φαρινάς είπε σε μια συνέντευξη πως η Κούβα είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πρέπει να τον βοηθήσουμε και αν τον βοηθήσουμε βοηθάμε όλους τους Κουβανούς. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε μόνους τους. Σας στείλουμε ένα μήνυμα μαζί με τους συναδέλφους μας πως ο κύριος Φαρινιάς έχει την στήριξή μας στον αγώνα του για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του κυρίου Γουγέρμου Φαρίνας και όλων των άλλων που αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κούβα. Συνεχίζουμε με την επόμενη υποψήφια που είναι η κυρία Μινέτου Χαϊντάρ. Την υποψηφιότητα έχει καταθέσει ο Νόρμπερ Νόιζερ, ο Βίλι Μάγερ, ο και, ε, Ρομέβα και η Ρουέντα και 40 Άλλου ευρωβουλευτέ. Πρώτα θα πάρει το λόγο ο κύριος Ρωμέβα η Ρουέντα και μετά ο Βίλι Μάγερ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τα ίδια λόγια του Ντάνι Κομπεντίτε. Πρόκειται για ένα αίσθημα που συμμεριζόμαστε απόλυτα ότι μία υποψηφιότητα δεν παρουσιάζεται κατά των άλλων υποψηφίων. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ε, υπερασπιστούμε την υποψηφιότητα της Αμινέτου Χαϊδάρ. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι η προσωπικότητα της υποψήφιας και οι λόγοι για τους οποίους ε, η αμινέ του Χαϊδάρ ε, ε, προχώρησε. Τώρα ακούγομαι καλά. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει όχι μόνο να τονίσουμε την προσωπικότητα της υποψήφιας αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν να στρατευθεί. Η αμυνέ του είναι γνωστή για την προάσπιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για το περιεχόμενο του μηνύματος που στέλνει αλλά και με τις μορφές τις οποίες το στέλνει. Εμείς ξέρουμε ότι για το βραβείο Ζαχάροφ ε, πρέπει να προωθούμε όλες τις απαντήσεις που δίνονται ε, στην αδικία που επικρατεί ε, στον πλανήτη. Η αμυνέ του πληρεί αυτό το χαρακτηριστικό, όχι μόνο λοιπόν προσωπικότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιστέκεται. Θεωρείται η, ο Σαχαριανή Γκάντι. Αυτό όμως που θα πρέπει να οδηγήσει την ε, Ευρώπη να αναλάβει ευθύνες είναι η εγκύτητα του χώρου στον οποίο προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα η αμυνέ του. Μέσα στα πλαίσια δηλαδή της ευρωμεσογειακής πολιτικής ε, και της ε, πολιτικής γυτνίασης, στο Μαρόκο παλεύει η του πρέπει να στείλουμε εμεί ένα μήνυμα ότι η καλή γειτονία με τις κοντινές μας χώρες δεν ε, σημαίνει ότι εμείς ε, αγνοούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπερασπιζόμαστε τα πιο θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι η Εμινέ του Χαϊδάρ ε, συγκεντρώνει όλες τις αξίες και τις αρχές του βραβείου Ζαχάροφ ξεπερνάει δε το μήνυμα στα όρια των ευρωμαροκοινών σχέσεων αλλά παίρνει τα όρια των ε, ευρωμεσογειακών σχέσεων. Ο Βίλι Μέγερ. Είναι ίσως αυτή μας η πρόταση, η μόνη πρόταση η οποία συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για, μια, ε, για ένα πρόσωπο το οποίο στρατεύεται στα πλαίσια της υπόθεσης και του αγώνα των Σαχαράουι. Είναι ίσως η τελευταία απικία, της, ευρωπαϊκή απικία της οποίας δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα και η, αποαπικιοποίηση η της Ερυθρέας ε, έγινε υπό την ευθύνη της Ισπανίας και το, χάος, και, και το πρόβλημα ε, η Ισπανία το έχει δημιουργήσει. Ο αγώνας των Σαχαράουι δεν περνάει καλές στιγμές. Η ίδια το απέδειξε όταν την απέλασαν από το, από το αεροδρόμιο του Λανθαρότε στην Ισπανία και ξεκίνησε την απεργία πείνας για να απαιτήσει κάτι το στοιχειώδες. Να σαν να γυρίσει στην Δυτική Σαχάρα. στο αεροδρόμιο της Ελ Αϊούν. Πάνω από 30 χρόνια γίνεται η συζήτηση για την αυτοδιάθεση της Ερυθρέας στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι η μόνη περίπτωση όπου η απαπικιοποίηση μία χώρα στην Αφρική ακόμη δεν έχει λήξει. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνονται σεβαστά τα δημοκρατικά δικαιώματα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης είναι κάτι το οποίο το έχουν εγγυθεί τα Ηνωμένα Έθνη ως βασικό δικαίωμα. Το βραβείο που θα δίναμε δεν θα ήταν ένα βραβείο προσωπικό προς την αμυνέ του Χαϊδάρη, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους τιμές. Θα έμεσα το βραβείο θα δινόταν στο λαό της Ερυθρέας και θα, έμεσα θα ήταν και μία πίεση προς τις μαροκινές αρχές που δεν του τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αυτή η απονομή θα ήταν ένα μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προς το Μαρόκο. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα της απεικιοκρατίας που πρέπει να λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέγερ. Ε, στον επόμενο υποψήφιο. Τον Ισάκ, ε, ε, τον οποίον προτείνουν ο Λεσμίτ, Σεσίλια Βίξτρομ, Μάριτ Πάλσεν, Ρένα Εκ και άλλοι 37. Να δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Λεσμίτ Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα ο Νταβίτ Ισακ είναι στη φυλακή 3.299 μέρες, σχεδόν πάνω από 9 χρόνια. 3.299 μέρες, πάνω από 9 χρόνια χωρίς δίκη, χωρίς καμία δίκη. Ο κύριος Ίζακ είναι Ερυθρέος δημοσιογράφος και θεωρώ πως έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη. Αλλά για εμένα το σημαντικότερο ε, όσον αφορά την εθνικότητά του είναι πως δείχνει την αφοσίωσή του στην ελευθερία του λόγου και του τύπου. Ο Ντάβιτ Ίσακ ζούσε ελεύθερος και ασφαλής στη Σουηδία αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Ερυθρέα για να ξεκινήσει την πρώτη ανεξάρτητη εφημερίδα αυτής της χώρας. Έλπιζε σε μια αλλαγή και σε ένα θετικό μέλλον της ε, χώρας του ένα μέλο στο οποίο θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ασκήσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και να μιλήσουν ελεύθερα. Θεμελιώδεις αξίες και για εμάς στην Ευρώπη. Δυστυχώς βεβαίω το όνειρό του δεν πραγματοποιήθηκε. Ανταυτού είναι στην φυλακή με το να φωτίσουμε το ζήτημα του Νταβίδη Ισακ θέλουμε επίσης να καταδείξουμε και την κατάσταση άλλων φυλακισμένων δημοσιογράφων που κρατούνται μαζί του χωρίς να έχουν κατηγορηθεί για τίποτα και χωρίς να έχουν περάσει δίκαιη δίκη. Κάτι το οποίο μας ανισχύει ιδιαίτερα καθώς ο αριθμό των πολιτικών κρατουμένων στην Ερυθρέα υπολογίζεται ε, στα 30.000 άτομα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το να δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ 2010 στον Ταβίτ Ίσακ δείχνει πως δεν αποδεχόμαστε τη μεταχείριση του κυρίου Ίσακ και των συγκρατούμενών του. Και πως μαχόμαστε για την ελευθερία του λόγου σε ολόκληρο τον κόσμο. Και θα ολοκληρώσω αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντας πως ο Νταβίτ Ίσακ μάλλον πεθαίνει στη φυλακή, ζει σε άθλιες συνθήκες Οπότε σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψηφίστε τον. Του χρόνου μπορεί να είναι αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Τώρα η κυρία Βίξτρομ. Έχετε τον λόγο. Δεν βλέπω την κυρία Βίξτρομ. Κύριε Σμιτ, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή αρκούν αυτά για τον υποψηφιό σας. Μου είπαν πως <clears throat> θα μιλήσει και η κυρία Βίξτρομ εκτός από σας για τον κύριο Νταβιδί Σακά, αλλά προφανώς λείπει. Οπότε να περάσουμε στον επόμενο υποψήφιο ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο. Με συγχωρείτε δεν με είχαν ενημερώσει κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Να το ξαναπώ όμως. <laughs> Ψηφίστε τον κύριο Ίσακ. Πεθαίνει στη φυλακή. Σας ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Επόμενος υποψήφιος, η επόμενη υποψήφιος είναι η κυρία Μπίρτουκαν Μιντέξα, την οποία προτείνουν ε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την παρουσίαση θα κάνει ο κύριος Άριαν Σέβεριν και η κυρία Γκόμες. Κύριε Σιδερίνη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι σοσιαλδημοκράτες και οι κύριοι αποφάσισαν να διαβοής να προτείνουν την κυρία Μπίρτουκαν Μιντέξα για το βραβείο Σαχάροφ του 2010. Η κυρία Μπίρτουκαν Μιντέξα είναι ηθίωπας πολιτικός η οποία το Δεκέμβριο του 2008 καταδικάστηκε σε ισόβια δεν μπόρεσε έτσι να είναι υποψήφια στις εκλογές του Μαΐου του 2010 παρά το ότι ήταν επικεφαλής της Ένωσης Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης. Η Διεθνής Αμνηστία την θεωρεί πολιτική κρατούμενο η οποία κινδυνεύει με βασανιστήρια μόνο και μόνο γιατί άρχισε ειρηνικά τα δικαιώματά της ε, ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεστε. Το δικαίωμα, το έγκλημα της ήταν το ότι μίλησε στην Σουηδία για το ότι αναγκάστηκε να υπογράψει για να της δοθεί χάρη το 2007 μαζί με άλλους 37 κρατούμενους οι οποίοι είχαν φυλακιστεί μετά από τις εκλογές του 2005. Η Μπίρτου Καρμιντέξα είχε πριν από αυτό συλληφθεί το Νοέμβριο του 2005 όταν το κόμμα της, ε, ο συναυσισμός για την ενότητα και τη δημοκρατία αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών. Οι εκλογές ήταν βίαιες και οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 187 άτομα δεν πυροβολήθηκε η κυρία Μύρη αλλά κατηγορήθηκε για προδοσία και καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Άνθρωποι που συνεργάζονταν με τους ε, κρατούμενους ε, κατέληξαν σε μια συμφωνία απονομής χάρης ε, και μαζί με άλλους 37 μετά από 18 μήνες φυλάκιση απελευθερώθηκε η κυρία Μπίρτου Καμιντέξα. Το Νοέμβριο του 2008 μίλησε σε μια δημόσια συγκέντρωση στην Σουηδία για την διαδικασία σύλληψη και απελευθερωσή της. Όταν επέστρεψε στην Αιθιοπία, οι αρχέ της ζήτησαν να ανακαλέσει τις δηλώσεις τη ή να συλληφθεί εκ νέου. Αρνήθηκε και συνελήφθη εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2008 όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακάλεσε την χάρη έκτοτε έχει μόνο σποραδική επαφή με δικηγόρους και η κατάσταση της υγείας της ε, χειροτερεύει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της Μπίτουκαν oh Μιντέξα σε ένα ψήφισμα μετά την σύλληψή της την δεύτερη φορά. Ο κύριος ε, Πίμπαλξ παραδέχτηκε το Μάρτιο του 2010 πως η φυλάξη της κυρίας Μιντέξα υποβαθμίζει την αξιοπιστία των εκλογών του Μαΐου του 2010, στην οποία το κυβερνών κόμμα κέρδισε ένα 99% των ψήφων και πιστεύω αυτό μιλάει από μόνο του. Το βραβείο Ζαχάροφ πρέπει να δίνεται σε αυτούς που χρειάζονται προστασία και διεθνή δημοσιότητα. Νομίζω πως η Μπύρ του θα τα χρειάζεται και τα δύο και στο πρόσωπό της βεβαίω θα εκπροσωπηθούν όλοι οι αιθίωπες πολιτικοί κρατούμενη, μία μητέρα όλας και μία από τις λίγες γυναίκες πολιτικούς ηγέτες στην Αφρική και θα δώσει δύναμη στους ξεχασμένους πολιτικούς κρατούμενους που αγωνίζονται για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Αιθιοπία. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες τώρα. Εγώ να προσθέσω στα όσα είπε ο κύριος Σεβερίν ότι Βεβαίως, τα όσα είπε για την Μπίρτουκαν ε, Τέξα δεν ε, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι αξίζουν λιγότερο, αλλά ε, συνάδελφοι, σας ρωτώ πόσοι την είχατε ακούσει αυτή τη γυναίκα, παρά το γεγονό ότι στην τελευταία θετία υιοθετήσαμε ψήφισμα που ζητούσε την απελευθέρωσή τη. Πρόκειται για μια νέα Αφρικανή γυναίκα, μια πολιτικό που αγωνίζεται για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στη χώρα τη και είναι επίσης μητέρα μικρών παιδιών. Τώρα που έχει πάλι κλειστεί στην φυλακή με ισόβιο κάθεξη, περνά μήνες στην απομένωση, χωρίς καμία επίσκεψη από για τους συγγενείς εκτός από τη μητέρα της και αγωνίζεται μέσα σε ένα ιδιαίτερα καταπιεστικό και ύπουλο καθεστώς. Ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί τη γλώσσα που εμείς στην Ευρώπη μας αρέσει να ακούμε, δηλαδή ανάπτυξη, δημοκρασία, ανθρώπινα δικαιώματα, που ενώ στην ουσία τα αρνείται στον κόσμο, στο λαό της. Όπως είπε ο Άντρεν Σεβερίν, Υπάρχουν χιλιάδε ε, πολιτικοί κρατούμενοι στην Αιθιοπία. Δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Η Voice of America και η Deutsche Welle είναι απαγορευμένε στην Αιθιοπία. Και μάλιστα καυχόνται που έχουν μπλοκάρει την Voice of America και την Deutsche Welle, ε, που έχουν μπλοκάρει τα blog και όλη την ε, επικοινωνία μέσω ίντερνετ. Εμείς είμαστε οι βασικοί δωρητές για αυτή τη χώρα, που είναι η δεύτερη πιο πολυκατοικημένη στην Αφρική. Και η Αφρικανική Ένωση έθελο τυφλή μπροστά σε αυτή τη χώρα. Είναι μια χώρα ακέ που έχει πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την ε, σύμβαση του Κοτονού. Γιατί κλείνουμε τα μάτια στα όσα συμβαίνουν. Είναι μια χώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει τίποτα όσον αφορά την υλοποίηση της διατησίας για τα σύνορα μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας που έχει αποτελέσει το αίτιο για τόσους πολέμους στην περιοχή είναι μια χώρα που εισέβαλε στη Σομαλία υπό την, την κυβέρνηση Μπούς υποτίθεται για να και μάλιστα υποστηρίζοντας τους ε, εξτρεμιστές, τους χαρσαμπάμ που αυτή τη στιγμή πολεμούν στη Σομαλία. Μα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις κυβερνήσεις μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να θελτυφλούν και γι' αυτό και σας ζητώ να στηρίξετε αυτή την υποψηφιότητα της ε, Μπίρτου Καρμιντέξα ώστε να στηρίξουμε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στην Αιθιοπία. Ερχόμαστε στον επόμενο υποψήφιο που είναι ο Πατήρ Θαντέος Νγκουέν Φανλή. Η υποψηφιότητα είναι από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ο κύριος Λαγκούτκο θα παρουσιάσει τον υποψήφιο. Του δύο τελευταίους υποψήφιους τυχαίνει να πρέπει να του παρουσιάσω εγώ και η υποψήφια αυτή δυστυχώ σχετίζεται με αυτό το λυπηρό γεγονό τη δίωξη χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρώτο υποψήφιο είναι ένα θαραλέο Ρωμαιοκαθολικό ιερέα από το Βιετνάμ είναι ο, ο πατέρας Γκυγέν Βαν Λί που γεννήθηκε το 1947 στο κεντρικό Βιετνάμ έγινε ιερέα το 1974 και ε, ε, διατέλεσε γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Γκουέν Κιμ Διέν. Χρησιμοποιεί τον αγώνα ανεβίας ως μέσο για να πετύχει τους στόχους του. Ο πατήρ Γουέν Βαν Λί υποστηρίζει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού Σε Ολόκληρη τη ζωή του έχει περάσει πάνω από 20 χρόνια στην φυλακή ή υποκατοίκον περιορισμό για την υποστήριξη ανθρωπίνων νόμων και τη δημοκρατία. Συνελήφθηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1977 επειδή με δύο δοκίμια του Αρχιεπισκόπου Γκουέν Κιμντίν, στα οποία επικρίνεται η καταπίεση των θρησκευτικών μειονοτήτων από την κυβέρνηση. Κατά την προσωρινή αποφυλάκησή του, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία τον Μάρτιο του 2010, ο πατήρ Γκουέν Φανλή τέθηκε αμέσως υποστενή επιτήρηση από τις αρχές και απειλήθηκε με σύλληψη πάσα στιγμή ως απειλή στην εθνική ασφάλεια επειδή ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να δώσει προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Ο πατήρ Γκουέν Φανλή συνοψίζει το έργο του για τη στήριξη των δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας ως εξής... Και παραθέτω, μια πολιτισμένη κοινωνία δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει σε καμιά κυβέρνηση, όποια και να είναι η ιδεολογία και οι πολιτικές αρχές της, να παρεκκλίνει από τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και να απομονώνει το λαό της πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα, επικαλούμενη τη μη ανάμεξη σε εσωτερικές κρατικές υποθέσεις. Τέλος της παράθεσης. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με διάφορους ε, ξένους ε, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ε, έκανε έκκληση στους συμπατριώτες του για μποϊκοτάρισμα του μονοκομματικού συστήματος διακυβέρνησης του Βιετνάμ, που είναι η ρίζα της θρησκευτική και πολιτικής καταπίεσης στο Βιετνάμ το μόνο ιδιωτικό τυπογραφείο του Βιετνάμ δημοσίευσε το Freedom of Speech, το οποίο είναι ένα φυλάδιο που συνέταξε ο πατέρας Γκέν Λί μαζί με άλλους τρεις ιερείς και διένυμε δωρεάν σε ολόκληρο το Βιετνάμ. Τον Μάρτιο όμως ε, έκλεισε αυτό το τυπογραφείο με παρουσία δικαστή, ε, εισαγγελέα, λόγω της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πατέρας Γκέν Βαν Λί ε, είναι φυλακισμένος πολλά χρόνια, ζει σε πολύ δύσκολες συνθήκες απομονωμένος και στερημένος από οποιοδήποτε πολιτικό δικαίωμα. Πάνω απ' όλα όμως ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε χάρη, υποτιθέμενη χάρη, που επιφυλάσσει το κομμουνιστικό καθεστώς στους Βιετναμέζους Ιερεί. Θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να μπορεί ο κόσμος να ζει με αξιοπρέπεια και ελευθερία. Έχει δείξει λοιπόν εξαιρετικό θάρρος ζητά ισότητα και δικαιοσύνη για τον λαό του και του Βιετνάμ και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Θα ήθελα να τονίσω πως ποτέ δεν έχει λάβει βραβείο Ζαχάροφ κάποιο πικός ε, του Βιετνάμ παρότι το Βιετνάμ είναι ένα καθεστώ με μια βίαιη κομμουνιστική δικτατορία πιστεύω πω ο πατήρ Νγκέν Βανλή αξίζει να λάβει το βραβείο αυτό και γι' αυτό σα ζητώ από όλου να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά του. Σα ευχαριστώ κύριε Λεγκούτκο. Ερχόμαστε στον τελευταίο υποψήφιο που είναι μια οργάνωση που ονομάζεται Open Doors, ανοιχτέ πόρτε και επίση προτείνεται από την Ευρω... Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και και πάλι ο κύριος Λεγκούτκο είναι εκείνος που θα παρουσιάσει την υποψηφιότητα αυτή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν τιμή μου και προνόμιό μου να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητα της οργάνωσης ε, της αποστολής Open Doors για το βραβείο Ζαχάροφ 2010. Είναι μια μη ομολογιακή χριστιανική αποστολή υποστήριξης των διοκόμενων χριστιανών. Παγκοσμίω, τρία τέταρτα των ανθρώπων που διώκονται για τις θρησκευτικές πεπιθήσεις είναι χριστιανοί. Σε διάφορους βαθμούς πραγματοποιούνται διώξει, διαφέρουν δηλαδή σε έντοση σε πολλές χώρες σαν τον κόσμο. Πρόκειται για μεμονωμένες πράξεις έω και οργανωμένη καταπίεση από τις αρχές. Η οργάνωση Open Doors ιδρύθηκε το 1995 από μια νεαρή Ολλανδέζα, την Άννα Βαντεμπέλ. Ύστερα από επίσκεψή της σε κομμουνιστικές χώρες όπως η δική μου, όπως όπου διώκονταν μάλλον χριστιανοί. Έφτασε στην Πολωνία και είδε ότι διώκονταν οι χριστιανοί εκεί και συγκινημένη από τον ε, κόσμο που συνάντησε και τις ιστορίες που άκουσε θεώρησε ότι έπρεπε κάτι να κάνει για να στηρίξει τον κόσμο αυτό. Όταν έφτασε πίσω στην Ολλανδία, η Άννα Βαντεμπέλ Έφτιαξε αυτόν τον οργάνωση που είναι γνωστή σήμερα ως Open Doors. Αρχικά στόχο είχε να φτάσει σε χριστιανούς στις κομμουνιστικές χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Σεχοσλοβακία και η Κίνα. Τη δεκαετία του 70 το πεδίο δράσης της επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή και σε τμήματα της Αφρικής αλλά και της Ανατολική... Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Επί του παρόντος η οργάνωση δραστηριοποιείται σε όλες... στις έξι πύρους και είναι δραστήρια σε πάνω από 50 χώρες όπου ε, καταπιέζονται ή διώκονται χριστιανοί. Άρα λοιπόν ε, αναπτύσσει δράση τόσο σε χώρες της Δύσης και σε χώρες με καταπιεστικά καθεστώτα για την προογή τη ελευθερία τη θρησκείας ή των πεπιθήσεων. Παρέχει νομική συνδρομή και στήριξη σε κρατούμενους και τι οικογένειέ του. Επιχορηγεί κέντρα αποκατάστασης για χριστιανούς πρόσφυγε, χείρε και παιδιά ε, διανέμει τη βίβλο και άλλα, άλλα χριστιανικά βιβλία. Αν και κάποιο από αυτή τη δουλειά πρέπει να γίνει με μυστικότητα, η Open Doors ποτέ δεν διστάζει να μιλήσει με τις αρχές και με όσους ε, έχουν πολιτικές θέσεις στις χώρες όπου λειτουργεί, ώστε να υποστηρίξει την ανοιξή θρησκεία. Η Άννα Βαντεμπέλ, για παράδειγμα, έχει μιλήσει με ηγε... κομμουνιστές ηγέτες στην Ανατολική Ευρώπη, με ηγέτες της Χαμάς στην Μέση Ανατολή και σήμερα μιλά με ηγέτες των Ταλιμπάν για να ζητήσει την συμφιλίωση. Να σας δώσω τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχήν έχουμε έναν ε, Ουσμπέκο Πάστορα, τον Δημήτρη, ο οποίος συνελήφθη το 2007 με κατηγορία παράνομης θρησκευτικής δραστηριότητας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Η Open Doors δημοσίευσε την ε, υπόθεσή του και εξασφάλισε ότι ο κόσμος δεν θα τον ξεχάσει. Ένα δεύτερο παράδειγμα Επίσης ε, η Open Doors ε, ε, υποστήριξε πακιστανικές ε, οργανώσεις χριστιανών που διώκονταν από τις πακιστανικές αρχές. Όλα αυτά τα χρόνια η Open Doors έχει στήσει γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει φτιάξει τον κατάλογο World Watch List, όπου κατατάσσει τις χώρες βάσει της ένταξης των διώξεων που υφίστανται για να τον κόσμο χριστιανοί επειδή ασκούν ενεργά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η Βόρειος Κορέα είναι η πρώτη στον κατάλογο, μετά είναι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. Ε, ε, στηρίζουμε αυτή την υποψηφιότητα. Η Open Doors είναι μια οργάνωση που δεν έχει καμιά άλλη φιλοδοξία από το να βοηθεί αλλήλους. Είναι μια οργάνωση που έχει φτάσει ξεπερνά μάλλον πολιτικές, ε, πολιτιστικά σύνορα, πολιτικά σύνορα, ενώ έχει ένα και μοναδικό στόχο. Μια αναποστολή να υπερασπιστεί την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία πίστης, ελευθερία συνείδησης, ελευθερία λόγου, ελευθερία του συναθρίζεστε και ούτω καθεξής. Η ελευθερία της πίστης είναι πολύ βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Εγώ πιστεύω πως η Open Doors αξίζει το βραβείο Ζαχάροφ για όλες τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά της στο παρελθόν, στα τελευταία δηλαδή 55 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεγκούτκο. Και τώρα συνάδελφοι ακούσαμε εννέα εξαιρετικούς υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάροφ Ελευθερία Σκέψης για το 2010 και είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι όλοι τους θα άξιζαν να πάρουν το βραβείο. Να κάνω μια ανακοίνωση πριν να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Ζολή. Φέτος το βραβείο Ζαχάροφ, ο Όλι Όλοφ, ο πρόεδρος του Memorial της Ρωσίας, έχει προσκληθεί στο Στρασβουργό ώστε να συμμετάσχει στην δημοσίευση, στην ανακοίνωση του υποψηφίου φέτος, στις 21 Οκτωβρίου. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι μας είπε πως δεν μπορεί καν δεν μπορεί να δεχτεί την πρόσκλησή μας, διότι Ο διοικητής της Τσετσενίας, Καντούροφ, του έχει ασκήσει ποινική δίωξη για συκοφαντία. Και πρόκειται να δικαστεί σύντομα. Το απαγορεύεται η έξοδος λοιπόν για τη Ρωσία. Είναι υποκατοίκον περιορισμών. Ε, από τη Ρωσία. Είναι υποκατοίκον περιορισμών. Ε, ας τους ευχηθούμε λοιπόν καλή τύχη και εκεί στη Ρωσία. Θα δώσω τώρα λοιπόν την προεδρία στη συνάδελφο Ζολή. Σα ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια σύντομη διαδικασία κάτσα 15 λεπτά δηλαδή για σας για να μπορέσετε να παρέμβετε και να πείτε τη γνώμη σας για τους υποψηφίους μας. Η κυρία Μουνίζ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω πως όλα οι υποψηφιότητες είναι βέβαια αξιοπροπείς, αλλά ωστόσο κάποιοι υποψήφοι αξίζουν το βραβείο περισσότερο από άλλους. Και αυτό για να ακουστεί η φωνή μας μέσω του βραβείου να ακουστεί η φωνή τους μέσω του βραβείου Ζαχάροφ εκείνων δηλαδή που δεν έχουν κάνει τα πρωτοσέλιδα των περιοδικών και των εφημερίδων. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι Υπάρχουν περιπτώσεις ε, με τις οποίες ασχολούμαστε μόνο σε συγκεκριμένες ε, φάσεις ενώ υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες άγγιξαν τη συνείδησή μας και ε, ακόμα και αν δεν έχουμε μπορέσει να κάνουμε κάτι για αυτούς. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε μία ευκαιρία σε εκείνους τους οποίους η γλώσσα τους θεωρείται διάλεκτος και η θρησκεία τους θεωρείται μία προκατάληψη και μόνο. εκείνους ε, που μπορούν να αποκτήσουν φωνή μόνο και μόνο μέσω αυτού του βραβείου. Να χρησιμοποιήσουμε το βραβείο για να είμαστε γενναιόδοροι, να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή σε εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι για να εξυπηρετήσουμε πολιτικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Donc, Σας ευχαριστώ για το πάθος με το οποίο υποστηρίζετε τους υποψηφίους σας. Είναι πολύ στιγματική στιγμή, πολύ έντονη στιγμή της κοινοβουλευτικής μας ζωής. Μπορούμε να διακρίνουμε, πρέπει να διαλέξουμε από έναν άνθρωπο που όλοι, αξίζουν, όλοι οι υποψήφοι αξίζουν το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σε μια οδυνηρή επιλογή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για όλα. Πρέπει να ορίσουμε ένα κατάλογο τριών υποψηφίων τη Δευτέρα το βράδυ 18 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Αυτό θα γίνει και κλεισμένο το θύρον. Και στη συνέχεια υπάρχει μια ψηφοφορία στην διάσκεψη των Προέδρων που επιλέγει τον υποψήφιο στις 21 Οκτωβρίου πάλι στο Στρασβούργο. Άρα η διάσκεψη των Προέδρων θα διαλέξει έναν και μόνο υποψήφιο. Το βραβείο μπορεί να απονεμηθεί τόσο σε ένα άνθρωπο, ένα άτομο ή σε κάποια οργάνωση που έχει νομική ε, οντότητα. 13 Δεκεμβρίου ε, ε, στο Στρασβούργο θα απονεμηθεί το βραβείο. Η τελετή 15 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στο Στρασβούργο. Όπως ήθιστε, η Γραμματεία του Ευρωκοινοβουλίου θα εξασφαλίσει την μάξιμουμ ε, διάδοση της δραστηριότητας. Εξάλλου προβλέπονται δραστηριότητες στο Στρασβούργο, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και στην πόλη του Στρασβούργου, στην ε, Χριστουγεννιάτικη αγορά. Η κυρία Βερζιά. Δύο λεπτά έχετε. Euh, Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, δεν ήθελα να παρέμβω για τις υποψηφιότητες αφού πήρα το λόγο, αλλά ήθελα να παρέμβω μετά από την ανακοίνωση που μας έκανε η κυρία Χάουταλα σε σχέση με το βραβείο γιατί αν δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε όταν ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βραβεύεται από το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο διότι υπόκειται σε καταστολή, ε, καταπίεση στη χώρα του, αυτό ξεπερνά τα πάντα. Δεν, σημαίνει τίποτα δηλαδή το να πονέμουμε ένα βραβείο Ζαχάροφ. Αν δεν είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τους δικού μας ε, βραβευθέντες, Μπορούμε να χτυπιόμαστε όσο θέλουμε, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει επίσημη διαμαρτυρία του Ευρωκοινοβουλίου κατά αυτού του λυπηρού γεγονότος, ώστε να επιμείνουμε απέναντι στις αρμόδιες αρχές, ώστε οι υπεύθυνοι του Μεμόριλα μπορούν να έρθουν τη στιγμή της απονομής του, γραφείου, του βραβείου Ζαχάροφ. Και δεν πρέπει να καταλήψουμε την προσπάθεια μέχρι τελευταία στιγμή. Ο κύριος Κονβεντήτ, ναι, να πω δύο λόγια. Είναι αλήθεια για το Memorial, αλλά ναι, καθεν ήταν αλήθεια για τα βραβεία Ζαχάροφ τη Κούβας. <coughs> το κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να βρει λύση. Δεν θυμάμαι όλους αυτούς που δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουν να πάρουν το βραβείο Ζαχάροφ. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για αυτού του είδους της χώρας. Και δεν μιλάω για τους ε, Ουζία που τους βάλανε στη φυλακή κατευθείαν. Ναι, ακριβώς εγώ για την Γκούτζα ήθελα να μιλήσω. Ούτζα και άλλους υποψήφιους. Βρεβευθέντες. Που ήταν στη φυλακή και εξακολουθούν να είναι στη φυλακή. Ούτζα, Άουν Σαντσουκί, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να ελευθερώσουμε κάποιους, όπως τον κύριο Σανάνα Λαγκούσμα, που είναι σήμερα πρωθυπουργό του Ανατολικού Τιμόρ, ε, τον ε, Λάσαν, που βγήκε από τη φυλακή και που μας είπε ο ίδιος πόσο πολύ μεγάλη διαφορά έκανε το βραβείο Ζαχάροφ για την προστασία του. Ναι, συμφωνώ με την κυρία Βεζιά ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε και να μην ξεχνάμε τους άλλους που είναι ακόμα στις ε, φυλακές. Και βεβαίως και οι ε, κουβανοί βεβαίως θα πρέπει να αναρτηθούν οι αφήσει τους εδώ μπροστά για να θυμίζουμε ότι ο αγώνας του συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω τον υποψήφιο από την Κούβα, αλλά αντιμετωπίζω το ίδιο δίλημα. Νομίζω πως οπωσδήποτε ο πρώτος ε, υποψήφιος εκπροσωπεί θύματα καταπίεσης αλλά ίσως να εκπληρώνει όλες τις συνθήκες. Συμφωνώ πως όλοι είναι άξιοι υποψήφοι, οπότε τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω πως ο αντίκτυπος που είχε στο παρελθόν το βραβείο Ζαχάροφ ήταν περιορισμένος. Γιατί αν δούμε τα διεθνή δίκτυα ε, πλην του Euronews δεν ασχολείται κανείς ούτε και ο τύπος. Ένα από τα μηνύματα λοιπόν που χρειάζεται να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα είναι πως ε, οι διπλωματικοί μας εκπρόσωποι στις χώρες ε, στις οποίες ζουν οι υποψήφοι και όσοι λάβουν το βραβείο θα πρέπει να είναι σε μόνιμη επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως του αν λάβουν το βραβείο είναι υποψήφοι. Και το όλο αυτό γιατί πρέπει να τονίσουμε όλους τους υποψήφιους. Η καλύτερη λύση θα είναι να δημοσιεύσουμε ένα αντιπροσωπευτικό βιβλίο Είναι φωτογραφίες, βιογραφίες και επιτεύγματα των διαφόρων υποψηφίων που δικαίως είναι υποψήφιοι όπως ακούσαμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να κρίνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να ψηφίσουμε έναν βεβαίως, αλλά αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να, να λύσουμε. Ευχαριστώ. Alors, euh, ναι, Είναι πραγματικά καταστροφικό το να διαπιστώνουμε ότι ο βραβευτής της περασμένης χρονιάς δεν μπορεί να παραβρεθεί στην ε, τελετή απονομής φέτος και με την Επιτροπή Διανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δούμε με ποια μορφή θα μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε. Θα εξετάσουμε την υπόθεση αυτή. Τελειώσαμε την συνεδρίαση μας, την κοινή μας συνεδρίαση. Συνεχίζει η συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. 18 Οκτωβρίου λοιπόν θα οριστεί ο κατάλογος των τριών επιλεγμένων υποψηφίων στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Πέρασε το τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν καθίστε. Ε, μπορείτε να βάλετε την καρτούλα στο σχετικό μηχάνημα. Σας παρακαλώ λοιπόν τώρα για πρακτικούς λόγους να ψηφίσουμε πρώτα τις γνωμοδοτήσεις και μετά θα ψηφίσουμε πρώτα λοιπόν τις νομοδοτήσεις, έκθεση Λίζεκ, υπέρ. για τις ε, θεωρήσεις ε, μεταξύ Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ, κατά. Α, μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία για την έκθεση Λίζεκ. Διευκόλυνση θεωρήσεων ε, 30 κάρτες είναι ε, στο μηχάνημα και 24 ψήφισαν. 24 υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάντα η έκθεση Λίζεκ, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την επανεισδοχή. ατόμων ε, από τη Γεωργία. 27 ψήφισαν. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 ψήφισαν 24 υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η Κόβατσεφ αρχίζει ψηφοφορία. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας 29 υπέρ 3 κατά και καμία αποχή. Ανθρώπινα δικαιώματα Έχουμε έναν κατάλογο για κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά στάνταρτ. Λοιπόν, συμβιβασμός 1, παράγραφος 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2, παράγραφος 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3, παράγραφος 1β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 6 δεν συμφωνείτε ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 5 αρχίζει ψηφοφορία Ναι, ναι, το έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίας με την προφορική τροπολογία. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία. 5 με την προφορική τροπολογία. Τριάντα τρεις υπέρ. Επτά κατά. Μηδέν εποχές. Οχτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Πρέπει να ψηφίσουμε και τη 12. Ωραία. 12. <coughs> υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 16 με, με την προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, έχω αμφιβολίες. Την ε, τροπολογία 19 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λοιπόν, 36 κατά και 8 υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία ονομαστική λοιπόν ψηφοφορία 50 κάρτες, 49 ψηφίσαντες, πέρας ψηφοφορίας, 49 υπέρ, ένας κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Bene, allora possiamo adesso procedere al punto riguardante il rafforzamento dell'OSCE e il ruolo dell'Unione Europea. Επόμενη έκθεση του κυρίου Ράουτσεκ που θέλει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα, συναδελφοί, στόχος του ψηφίσματος είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τον ρόλο του ΟΑΣΕ και βεβαίως ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πριν από την Σύνοδο. Είμαστε σε μια εποχή μετά την Λισαβόνα, οπότε έχει λόγο μεγαλύτερο το κοινοβούλιο μας, οπότε στόχος μου ήταν να μιλήσει με μία φωνή στη Σύνοδο Κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν συζητήσαμε αυτό το ψήφισμα αρχές Σεπτεμβρίου σας ζήτησα να συνεισφέρετε με ιδέες σε αυτό το ψήφισμα, το κάνατε. 140 συνολικά τροπολογίες, οφείλω να πω πως περισσότερες ήταν πολύ επικοδομητικές, εμπλούτησαν το ψήφισμα. Μαζί με τους κοιόδης εισηγητές προσπαθήσαμε να τις βάλουμε σε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες και φτιάξαμε 8 τον αριθμό, τις οποίες ελπίζω όλοι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ λοιπόν για την συνεισφορά σας. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, να ευχαριστήσω κάποιους όπως τον κύριο Σόλτς, ο οποίος απέσυρε κάποιες τροπολογίες και ελπίζω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να έχουμε μία φωνή ολόκληρης Επιτροπής Εξωτερικών και σε δύο εβδομάδες βεβαίως του Κοινοβουλίου ολόκληρου για να κληρώσουμε έτσι αυτό τον ρόλο του Κοινοβουλίου να μιλάει με μία φωνή και με δυνατή φωνή να μιλήσει με δυνατή φωνή στην Σύνοδο Κορυφή στην Αστάνα. Ευχαριστώ κύριε Ρούτσεκ. Συγγνώμη Ρόιτσεκ, συγγνώμη για την λάθος ε, προφορά του ονόματός σας πριν. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε από την τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν συμφωνείτε. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 18. 44-45 non sono ancora tutte, però insomma 47. Λοιπόν, από ε, τις, από τις 52 κάρτες έχουν ψηφίσει 48 πέρα στις ψηφοφορίες 21-26. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε το συμβιβασμό 1. Θα το ψηφίσουμε σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπάρχει μία τροπολογία που προτείνει ο κύριος Ζιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα μεταξύ του refusal και των NATO member states να υπάρξει μία αλλαγή και να τη διαβάσω αγγλικά η συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Bene, allora non ci sono opposizioni a questo emendamento orale. σε αυτήν την προφορική τροπολογία. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα κύριε Πρόεδρε. Votiamo l'emendamento orale. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία που μόλις μας ανέφερε ο κύριος Ζιπ και που αφορά στο δεύτερο τμήμα του συμβιβασμού 2. Και προσθέτει μέχρι τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτός ο συμβιβασμός, με αυτόν τον συμβιβασμό πάμε στο συμβιβασμό 4, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 36 34, 34, με συγχωρείτε. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει, διότι έχουμε εγκρίνει το συμβιβασμό 1 και το τρίτο τμήμα της τροπολογίας 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αποσύρθηκε 37 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42. Τις... Ψηφίζουμε τη 41 γιατί αποσύρθηκε 37. Υπέρ τη 41. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. <coughs> Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 42. Ωραία. Να, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 42. «53 κάρτες ψήφισαν και οι 53 κάρτες, πέρας ψηφοφορίες, 25 υπέρ, 28 κατά. Δίκιο είχατε. Απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές δεν μου φαίνεται σαφές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 46 αρχίζει η ψηφοφορία 52 ψηφίσαντες. 29-23 εγκρίνεται. 40... Σαράντα εφτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σαράντα οχτώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 με την προφορική τροπολογία του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, 56 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβασμός, απορρίπτεται, συμβιβασμός 2. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονικός έλεγχος για την 59. 53 κάρτες. 53 ψηφίσαντες, 21-32 το σκορ απορρίπτεται. 63. Προφορική τροπολογία του κυρίου Κυριλόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο προτείνω είναι στο τέλος της παραγράφου 13 που τελειώνει in the impact of population movement κτλ. να προσθεθεί συμπεριλαμβανομένων ε, including that of IDPs and refugees, γιατί ξέρουν πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα άτομα αυτά και στα Δυτικά Βαλκάνια και στο Νότιο ε, και, στη, και στην Κυργυζία. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Στο τέλος της παραγράφου including that of ADPs and refugees, να προσθεθεί. Il relatore ha fatto conoscere con il linguaggio del corpo che è d'accordo. Ο εισηγητής έγνευσε ότι συμφωνεί. Συμφωνώ, συμφωνώ λέει ο εισηγητής και προφορικά. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 71 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα της 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 71 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Ε, εντάξει. Ψηφίζουμε ελληνικά λοιπόν για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 71. Άρχεται η ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος των σοσιαλιστών. Τέλος της ψηφοφορίας, 53 ψήφισαν, 23 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τη τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε. 71 τρίτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. «53 ψήφισαν, όχι, 53 έβαλαν την κάρτα, 52 ψήφισαν. 26 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Προφορική τροπολογία του κύριου Τζίπε. Που μπορεί να μας πει ποια είναι. Παρακαλώ κύριε Τζίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρότασή μου είναι να αντικατασταθεί η αγγλική λέξη appropriate από ε, important. Το σημαντικό φόρουμ για να συζητηθούν αυτό το είδος οι προτάσεις. Και το δεύτερο τμήμα προτείνω η παράθεση 7, η αιτιολογική σκέψη 7 να να το τελειώσει με τις λέξεις Νοέμβριο 2008. Tutte e due, sì. Quindi anno importa e poi la, eh, si esclude 2009. Eh, Finire, 2009. Finire col 2009 si esclude il resto. Τι να λέει με το 2009, να τελειώσει το 2009 και να απομει... τα υπόλοιπα να διαγραφούν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρόταση του κύριου Γκζίμπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 7 εγκρίθηκε λοιπόν και πάμε έτσι στην τροπολογία 81 όπου υπάρχει μια άλλη προφορική τροπολογία. Ο πρωταγωνιστής της συνεδρίασής μας σήμερα είναι ο κύριος Ξύμπ. Μπορείτε να μας πείτε τι θέλετε εδώ, την προφορική σας τροπολογία. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρότασή μου είναι να προσθέσουμε μετά τη λέξη ε, Ρωσική Ομοσπονδία και τη λέξη Ουκρανία να προσθεθεί ΙΠΑ και ΝΑΤΟ. Κύριος Ράουτζικ. όχι είμαι κατά, γιατί είμαι κατά ολόκληρες τροπολογίες. Δεν έχει νόημα να είμαι υπέρ αυτών των, ε, αυτής της προσθήκης, αφού είμαι υπέρ ολόκληρες τροπολογίες. Bene, eh, Οπότε προτείνω να κάνουμε χωρί δύο χωριστέ ψηφοφορίε για την τροπολογία 81. Η πρώτη είναι το κείμενο όπω ήταν προηγουμένω, πριν δηλαδή να παρέμβει ο κύριο Γκζίμ. Αν εγκριθεί. Εντάξει. Αν όχι, Παρακαλώ κύριε Γκάλερ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως η προφορική τροπολογία του συναδέλφου Ζιπ έχει... θα είχε νόημα εάν είχε πιθανότητα να περάσει η τροπολογία, αλλά έχουν εντύπωση πως εάν οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ είναι κατά της τροπολογίας, ε, δεν χρειάζεται καν η προφορική τροπολογία. Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di questo... Έτσι έχουν τα πράγματα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για την 81. Λυπάμαι. Κύριε Ξέπ. Υπέρ της 81. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ωραία αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 δύο τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 84. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 84 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ του δεύτερου τμήματος της 86 κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι βέβαιος ας το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να δούμε για την 91 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Πέντε σε ψήφισαν. 26 κατά, 25 υπέρ. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Να ελέγξουμε και για την 93 παρακαλώ. Ελεκτρονικός έλεγχος για την 93. 32 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται θα έλεγα. 97 υπέρ. Κατά αποχές δεν είμαι βέβαιος. Θα έλεγα με το μάτι ότι είναι υπέρ, ότι εγκρίνεται δηλαδή. Αλλά δεν τα σηκώνετε όλα τα χέρια σας. Όχι, πάμε στην 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Άμα θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Αλλά εγώ θεώρησα, είδα ότι απορρίφθηκε. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Όχι, όχι, να διορθώσω μισό λεπτό. Πρέπει να ψηφίσουμε την 10 γιατί η 9 δεν εγκρίθηκε. Άρα, για τη 10 να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, επίση απορρίψαμε την 7, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε και για την 8. Υπέρ τη 8. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Τι θέλετε, οι σοσιαλιστές ζητούν ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. 56, 56 ψηφίσαντες, 29 κατά, 27 υπέρ, απορρίπτεται. 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, ήταν η 4 τώρα υπέρ κατά αποχές. Εδώ δεν είμαι βέβαιος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 4 ηλεκτρονικά. 55 ψήφισαν, 27 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο της ε, έκθεσης όπως τοποποιήθηκε. Σας κάνω αναμετάδοση. Λοιπόν, 56 κάρτες έχουν τοποθετηθεί στις σχισμές, 56 εψήφισαν, 49 υπέρ, μία κατά, 6 αποχές. Μπράβο σας, κύριε Σιγητά. Συγχαρητήρια. Allora, grazie. Ωραία. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών για την ε, δουλειά που έκανε. Τέλος τώρα και αρχίζει το διευρυμένο Προεδρείο μόλις θα έχει αδειάσει η αίθουσα. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ.